No, I don't want them, but... Good, evening, colleagues. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Καλώς ορίζω τα μέλη των Επιτροπών Έκων και Λίμπη. Αρχίζουμε. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, την ημερήσια διάταξη εγκρίνεται γλωσσικό προφίλ. Δυστυχώς, γκέλικ δεν θα έχουμε. Και θα μειωθούμε στις 16 γλώσσες από τις 7 ε, μέχρι τις 8. Η ψηφοφορία θα είναι σε 7,5 αν έχετε τις κάρτες. Αυτά από τη δική μου την πλευρά. Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΟΝ θα συνεχίσει για 10 λεπτά, ενώ εγώ μίλησα τόσο λίγο. Λοιπόν, Πέταρ, εσύ. Να καλωσορίσουμε πρώτα την Επίτροπο Γιούροβα που είναι αρμόδια για δικαιοσύνη καταναλωτές και ισότητα των φύλων και θα συζητήσει με τις δύο επιτροπές αφού συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τους συντονιστές. Ευχαριστούμε που ήρθατε ανανεωμένοι. Στις 27 Οκτωβρίου υπάρχει καινούρια κατεξοδότηση πράξη σχετικά με υψηλού κινδύνου τρίτες χώρες που έχουν προβλήματα κατά πολέμηση τρομοκρατίας και ξέπλυμα χρήματος. Το Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο και τον Μάιο φέτος είχε κάποιες αντιρρήσεις. Θα πρέπει να γίνει καλός διάλογος με την Κομισιόν, να δούμε πόσο τριμερής διάλογος και η πέμπτη οδηγία για το ξέπλυμα του χρήματος θα συνεχιστεί και θα προχωρήσει. Εμείς ε, θέλουμε να παραταθεί μέχρι 27 Δεκεμβρίου, κατά ένα μήνα δηλαδή, η προθεσμία. Αυτή είναι καλή ευκαιρία για να συζητήσουμε για το δικό χάρτη, για το πώς θα προχωρήσουμε, που έχει τίτλο «Προς νέα μεθοδολογία για την αξιολόγηση της Ένωσης των χωρών υψηλού κινδύνου» και την ε, οδηγία του 2015 για την ε, καταπολέμηση ξεπλήματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Πήραμε τον οδικό χάρτη μετά τη δεύτερη ένσταση του Κοινοβουλίου με βάση την πολιτική δέσμευση της Επιτρόπου. Η Κομισιόν τώρα εξετάζει ποια μεθοδολογία θα είναι πλέον ενδεδειγμένη για την αξιολόγηση των τρίτων χωρών από την πλευρά της και Προσβλέπουμε να ακούσουμε από την Επίτροπο τι τελευταίες εξελίξεις. Και μέσα από το δικό σας πρίσμα θέλω να σας ζητήσω να μας δώσετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για την βιωσιμότητα της εφαρμογής μιας τέτοιας μεθοδολογίας σε έφθετο χρόνο σύμφωνα με το δικό χάρτη ειδικότερα. Όπως συζητήθηκε με το επιτελείο σας προηγούμενη εβδομάδα, θέλουμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε πιο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για τη νέα μεθοδολογία. Δεύτερον, σας ζητώ επίσης να δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία, ειδικότερα σχετικά με την ε, διαφάνεια σε σχέση με την πραγματική ιδιοκτησία που αναφέρει η Κομισιόν ως ένα κριτήριο στον οδικό χάρτη που μπορεί να συμπεριληφθεί. Η, νέα, η νέα μεθοδολογία ακολουθεί το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας αυτόνομης αξιολόγησης από την Κομισιόν των Τρίτων Χωρών που θα μπαίνουν στον κατάλογο. Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι χρησιμοποιώντας την, τον κατάλογο FATF της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι. Ενώ το AMLCTF, αυτέ αυτές οι αδυναμίες μπορεί να επιμένουν στις χώρες αυτές εις ό,τι αφορά διάφορες πτυχές που καταγράφονται στο άρθρο 9. Έχουμε καταγράψει κάποια αποτελέσματα της συνεχιζόμενης αυτής εργασίας, ειδικότερα σχετικά με την απόφαση της Κομισιόν να διατηρήσει τον κατάλογο όλες τις χώρες που προηγουμένως είχαν συμπεριληφθεί παρόλο που ακόμα δεν είναι στην AFTF, ε, ε, Ουιάννα, Λαρμπιριάρ και Αφγανιστάν ε, για να διαγραφούν από τον κατάλογο χώρες αυτές η Κομισιόν πιστεύει ότι χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση για να ελέγξουμε τις προόδους των χωρών σε σχέση με τις στρατηγικές τους αδυναμίες. Γι' αυτό παράλληλα με αυτή την αρχή της προφύλαξης ε, ε, χρειάζεται δέουσα επιμέλεια περισσότερο στη Γουιάννα, Λαού και το Αφγανιστάν. Επίσης, ε, σημειώσαμε και το νέο σχέδιο πράξης που δόθηκε για διαβουλεύσεις στην ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών και που στηρίζεται στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες μετά τη συνάντηση του Νοεμβρίου του FATF. Σε σχέση με την Αιθιοπία θεωρούμε ότι η επόμενη κατεξουσιοδότηση πράξη θα βάλει Σρι Λάγκα, Τριντάν και τον Πάγο και την Ισία στις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου της Ένωσης. Αυτό αναφέρεται στη γνώμη της Κομισιόν ότι χρειάζεται να εκδίδονται κατά εξουσιοδότηση πράξης ούτως ώστε να βεβαιωνόμαστε ότι οι κανόνες της Ένωσης θα ισχύουν στις τρίτες χώρες που διεθνώς θεωρούνται ό,τι είναι υψηλού κινδύνου. Μετά από αυτή τη μακρά, πολύ μακρά εισαγωγή που δίνει το πλαίσιο, αρχίζουμε τη συζήτηση. Θα προεδρεύσει ο πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Σας ευχαριστώ πολύ Πέτερ. Ευχαριστώ την Επιτροπή ΕΚΟΝ και την Γραμματεία. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία για το θέμα αυτό. Να σας υπενθυμίσω και εγώ ότι το Κοινοβούλιο υπέβαλε δύο ενστάσεις ε, Ιανουάριο και Μάιο για την κατεξοδότηση αυτή πράξη και η Κομισιόν επανειλημμένω έχει πει ότι είναι ξεκάθαρο ότι στη συνάντηση που είχαμε την Τρίτη στην κοινή συνεδρίαση έγινε μια ανταλλαγή απόψε για την πρόοδο και για τη μεθοδολογία. Καλό είναι όμως να ακούσει όλη η Επιτροπή Λίμπε και όλη η Επιτροπή ΕΚΟΝ τι έχει να πει επίτροπος σε σχέση με την πρόταση του Μαΐου και τη μεθοδολογία και τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε. Τα είπε και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Θα καλέσω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου την Επιτροπή Γιούροβα να πάρει το λόγο για 10 λεπτά, να κάνει την ε, δήλωσή της και εφόσον υπάρχουν ερωτήσεις σχόλια θα ακολουθήσει ένας γύρος ανταλλαγής απόψεων με τα μέλη των δύο επιτροπών. Κυρία Γιούροβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι, αξιότιμοι βουλευτές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ προσωπικά για να σας ενημερώσω για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, συγκρότηση ενό αυτόνομου ενωσιακού καταλόγου τρίτων χωρών που παρουσιάζουν υψηλό ε, κίνδυνο για το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Ζητώ συγγνώμη ε, για την απουσία της προηγούμενης εβδομάδος γιατί πιστέψτε με, το να μην μπορεί ένα πολιτικό να ανοίξει το στόμα του και να πρέπει μόνο να ακούει γιατί χάσει τη φωνή του είναι καταστροφή. Και ευχαριστώ για την κατανόησή σα. Η Επιτροπή Πάνα συζήτησε τη σημασία τη καταπολέμηση του ξελίματο χρήματο την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ πρέπει να περιλάβουμε ένα φιλόδοξο ενωσιακό πλαίσιο κατά χωρών και δικαιοδοσίων που δεν σέβονται του κανόνε της ε, ε, καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Έχω ακούσει αυτό που λέτε, ότι πρέπει να εντοπίσουμε με ένα νέο σύστημα της χώρας ψηλού κινδύνου και να έχουμε ένα εύρωστο ε, και νομικό στέρεο σύστημα. Με αυτό θα στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υψηλά πρότυπα για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού εγκλήματος. Πρότυπα που καθιστούν δύσκολο για εγκληματίε και φοροαποφεύγοντες να εκμεταλλεύονται πολύ απλά τον παγκόσμιο χαρακτήρα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όταν συνδεθήκαμε τον Ιούλιο, σας ε, παρουσίασα ε, σε αδρές γραμμές ε, τη μεθοδολογία μας για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου και τώρα είμαι εδώ για να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς εμείς σκοπεύουμε να προβούμε στην δική μας εξολόγηση και να λάβουμε υπόψη και τη δική σας συμβολή. Καταρχάς, πώς θα εντοπίζονται οι χώρες προτεραιότητας που πρέπει πρώτα να αναλυθούν ξέροντας ότι δεν μπορούμε βέβαια να εξολογήσουμε 200 χώρες με μιας. Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που μου θέσατε, άλλωστε και τον Ιούλιο στη συνάντησή μας. Μετά θα σας μιλήσω για τα κριτήρια που προθέμενα να χρησιμοποιήσουμε, λαμβάνοντα υπόψη ότι η αναθεώρηση τη οδηγία για την καταπολέμηση τη ομοποίηση των παραγωγών δραστηριότητε, ξέπλυμα χρήματο, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, δυστυχώ. Έπειτα θα μιλήσω για την πρότασή μας. Δηλαδή, τι θα κάνουμε μέχρι την, πρώτη, ε, την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Για το πρώτο ζήτημα, θεωρώ ότι η διαδικασία της καταγραφής αυτής πρέπει να είναι ένα εργαλείο για στοχευμένη αποτελεσματική αποδοτική πολιτική της Ένωσης ε, κατά χωρών υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, η Κομισιόν θα πρέπει να μπορεί να εντοπίζει για ποιες χώρες θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αξιολόγηση και κατά πρώτον θα πρέπει να εντοπίσουμε τις χώρες που είναι πιο σημαντικές και πρέπει να αναλυθούν. Αφετηρία για αυτόν τον κατάλογο της Ένωσης θα είναι το έργο της ομάδος χρηματοοικονομικής δράσης, που πλήρες μέλος της είναι και η Κομισιόν. Οι χώρες οι οποίες ε, αποτελούν κίνδυνο για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα θα ε, πρέπει να θεωρούμε ότι είναι εξίσου επικίνδυνε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο στόχο του καταλόγου. Υπάρχουν κάποιε χώρε βέβαια που δεν έχουν ε, αναγνωριστεί ω επικίνδυνε από την ομάδα χρηματοοικονομική δράση, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα πρέπει κάπω να αντικαθρεπτίζεται στην πρότασή μα. Προτείνουμε λοιπόν να εστιάσουμε σε ορισμένε από αυτέ τι 200 δικαιοδοσίε σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση τα εξή κριτήρια. Πρώτον, οι τρίτες χώρες οικονομικής συνάφειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μείζωνα χρηματοπιστωτικά κέντρα και οι χώρες με στενούς οικονομικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα λαμβάνουμε υπόψη τις χώρες εκείνες οι οποίες ε, είναι στο πλαίσιο του screening ε, του καταλόγου που ο συνάδελφος Μοσκοβισή επεξεργάζεται μαζί με τα κράτη-μέλη. Μιλάω για τον τομέα της φορολογίας αυτός ο κατάλογος, το screening αυτό θα ολοκληρωθεί ήδη την εβδομάδα αυτή. Δεύτερο κριτήριο. Τρίτε χώρε οι οποίε έχουν εντοπιστεί από την Europol και την Ευρωπαϊκή Μέση Εξωτερικής Δράση, χώρε οι οποίε παρουσιάζουν κινδύνους ε, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τη Δημοκρατία και τις νομοσπιστής των παράνομες Έτσι θα καλύψουμε και με τον εντοπισμό τρίτων χωρών όλε τι χώρε. και αυτέ που δεν τις έχει στην κατάλογο της και τι τις εξετάζει η ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης. Δεν θέλουμε να έχουμε τυφλά σημεία. Οποιαδήποτε δηλαδή χρονική στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να επεκτείνει το πεδίο και να καλύψει προς τρεις χώρες, ανάλογα παραδείγματο χάρη, με νέα στοιχεία ή σε συνάρτηση με νέες πληροφορίες ε, που θα ε, ληφθούν. Στο δεύτερο στάδιο θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες, τη σειρά προτεραιότητες με, με την οποία θα αξιολογούμε τις δυνητικά επικίνδυνε χώρες. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα εξή κριτήρια προτεραιότητα σε αυτή τη φάση. Πρώτον, τρίτε χώρε που είναι ε, στον ε, ενωσιακό κατάλογο των ε, χωρών ή που δεν συνεργάζονται. Αυτό το εγχείρημα είναι σε εξέλιξη από τον Επίτροπο Μοσκοβισή και θα καταλήξει σύντομα. Δεύτερον, τρίτες χώρες για τις οποίες ήδη έχουμε υλικό στη διάθεσή μας που να στηρίζει την αξιολόγησή μας. Χώρες δηλαδή που ήδη έχουν αξιολογηθεί από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης στο πλαίσιο του Νοδικού Χάρτη. Τρίτον, τρίτες χώρες που έχουν ήδη επισημανθεί ως εκτεθειμένες σε εγκληματικέ δραστηριότητες ή τρομακρατικές απειλές. Στην προκειμένη περίπτωση, οι πληροφορίες της Europol ή της ΕΙΕΔ έχουν μεγάλη σημασία. Τέταρτον, τρίτες χώρες που πρόσφατα βγήκαν από τον κατάλογο της ε, ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης η ράξη των προτεραιοτήτων εδώ θα δικαιολογείται από το γεγονός ότι αυτή η απαλληφή από τον κατάλογο ε, θα μελετάτε για να δούμε κατά πόσο είναι επαρκή τα στοιχεία και δικαιολογούν την απαλληφή από τον κατάλογο. Αυτό είναι άλλωστε αυτό που κάνουμε ήδη με τις χώρες που προτείνονται για αυτό το delisting. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Το τρίτο στη μεθοδολογία. Θέλουμε να ορίσουμε κριτήρια για την αξιολόγηση του κινδύνου. Η νομική βάση για αυτή την αξιολόγηση στηρίζεται στο άρθρο 9 της οδηγίας για το ξέπλυμα του χρήματος που σήμερα έχει στοιχεία όπως ποινικοποίηση του ξεπλήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, προϋπόθεση, ε, ε υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών. Θέλουμε να επεκτείνουμε τα κριτήρια όμως στα πλαίσια της αναθεώρησης της οδηγίας να βάλουμε στοιχεία όπως αποτελεσματικότητα των κυρώσεων και διεθνή συνεργασία. Η Προεδρία εξέτασε και θα δώσει συνέχεια τον επόμενη εβδομάδα στον τριμερή διάλογο στα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν θα εξετάσει ως ε, βασικό κριτήριο την πραγματική ιδιοκτησία που πρέπει να ε, υπάρχει. Επιμένω ότι θα ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει πλέον ανοχή σε δικαιοδοσίες που χρησιμοποιούν ή διευκολύνουν ε, αδιαφανείς δομές. Αυτά έχουν τελειώσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα. Εδώ θα πρέπει να προχωρήσει περισσότερα, περισσότερο από ότι G8, G20 ε, ή η ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης, η FATF. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης θα υπάρχουν τέλος του 2018 για την πρώτη ομάδα των, ομάδων, των χωρών προτεραιότητας. Η αξιολόγηση άλλων σημαντικών χωρών θα αρχίσει αμέσως σε ένα δεύτερο στάδιο μετά το 2020. Για τη δεύτερη ομάδα χωρών θα κάνουμε σταδιακά τις εργασίες μας στο βαθμό που θα έχουμε νέες πηγές πληροφοριών ή κατεπήγοντα θέματα. Για παράδειγμα, νέες ε, εκθέσεις αξιολόγησης. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να προσθέτουμε σταδιακά χώρες στον κατάλογο μετά το 2019. Αυτό σημαίνει παράλληλα ότι δεν θα περιμένουμε μέχρι το 2025 για να ολοκληρώσουμε όλο τον κατάλογο Συνεχώς θα προσθέτουμε χώρες στο μεσοδιάστημα. Για το δεύτερο κύμα χωρών έχουμε λιγότερες πληροφορίες και λιγότερες ανησυχίες και διακυβεύματα εκτός αν υπάρχουν απρόβλεπτα. Είμαι πρόθυμη να σκεφτώ να εισαγάγουμε ε, ε, κάποια απρόβλεπτα και κατεπήγοντα προβλήματα. Τότε θα εξετάζει κατεπήγοντος και η Κομισιόν αυτές τις χώρες και θα ε, εντοπίζει τυχόν ανεπάρκειες. Εν τω μεταξύ η Κομισιόν θα παρακολουθεί τις χώρες που αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο, θα παρακολουθεί την πρόοδο και αν ε, δικαίως αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο μπορεί να αφαιρεθούν και άλλες. Ε, αυτά είναι τα στάδια της μεθοδολογίας. Οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών θα συμμετέχουν στην ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων για το ξέπλυμα και την τρομοκρατία που επικουρεί την Κομισιόν όταν προετοιμάζει κατά εξουσιοδότηση συμπράξεις. Το Ευρω... Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καλούνται σε κάθε συνεδρίαση. Η επόμενη θα γίνει με ειδικού ε- εθνικούς εμπειρογνώμονε στις 11 Δεκεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει το ίδιο υλικό και τις ίδιες πληροφορίες όπως τα κράτη-μέλη. Πρέπει να εργαζόμεθα με τρόπο διαφανή. Η διαφάνεια ε, οδηγεί σε εμπιστοσύνη στη διαδικασία, ε, εμπιστοσύνη και στα αποτελέσματα. Η διαφάνεια επίσης ε, διασφαλίζει ότι οι ανεπαρκείς τρίτες χώρες θα ξέρουν τις προσδοκίες μας και θα βελτιώνουν τις αδυναμίες τους. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να κάνει αναφορά στο Κοινοβούλιο όσο συχνά ε, χρειάζεται και στο Συμβούλιο. Είναι σημαντικό η μεθοδολογία αυτή να ε, ολοκληρωθεί ε, στα πλαίσια των δύο επιτροπών. Συμφωνούμε ότι η δημιουργία ενός σταθερού καταλόγου σίγουρα θα διευκολύνει το έργο μας. Θα πρέπει να έχουμε και τους απαραίτητους πόρους ε, και τους ε, ε, δημιουργούμε τώρα. Ευχαριστώ που μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τέλος, για την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης. Το... Η ανεξάρτητη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ωφελήσει πάρα πολύ την Κομισιόν. Αυτές οι αναλύσεις θα αυξήσουν την ε, κατανόησή μας των κινδύνων των χωρών και θα βελτιώσει την ενισχυμένη μας παρουσία στην ε, ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης, ε, ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των ανεπαρκειών των τρίτων χωρών. Θυμίζω ότι συνεχίζω να πιστεύω ότι η ΦΑΤΦΗ, η ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης, είναι πολύ σημαντική, πρέπει να την υποστηρίξουμε και θα πρέπει να δουλέψουμε στρατηγικά και πολιτικά στις συζητήσεις που γίνονται σε αυτό το φορέα. Η Κομισιόν ήδη έχει αυξήσει σημαντικά την εμπλοκή της στην ε, ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης. Είναι αναπόφευκτο να έχουμε και μια ενδιάμεση περίοδο μέχρι να πάρουμε τα πρώτα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή της νέας ε, μεθοδολογίας μέχρι το τέλος του 2018. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Το να κάνουμε τίποτα δεν είναι επιλογή στο διάστημα αυτό. Η Κομισιόν έχει νομική υποχρέωση να ε, ε, εκδώσει κατεξουσιοδότηση πράξης ώστε να ε, εντοπίζονται οι χώρες υψηλού κινδύνου. Μέσω ότου ολοκληρώσει την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της μεθοδολογίας οτιδήποτε άλλο θα αποτελούσε ανευθυνότητα, λαμβάνοντα υπόψη το επίπεδο τη ολοκληρώση των χρηματοστατικών συστημάτων, την εσωτερική αγορά που θα εξετίθεται σε σοβαρού κινδύνου ξεπλήματο χρήματο και τρομοκρατία, χρηματοδοτήση των τρομοκρατών, αν δεν έχει. Ε, αν δεν βάλουμε στην, αυτά που έχει εντοπίσει η ΦΑΤΦ στη δικαιοδοσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, δεν θα συμμορφωθεί με τη διεθνή υποχρέωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι δεν θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την παγκόσμια προσέγγιση προς τις χώρες υψηλού κινδύνου. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να υποστηρίξετε την κατεξοδότηση πράξη που σας έχει υποβληθεί προς εξέταση. Έχουμε λήψει στρατηγικές όσον αφορά το καθεστώς για το ξέπλυμα χρήματος. Και το κέρας της Αφρικής είναι ευαίσθητη περιοχή όσον αφορά την δρομοκρατία. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη, Αυτά είναι τα προκατακτικά που έχω να πω, αυτές είναι οι σκέψεις μας. Είμαι εδώ για να ακούσω ανησυχίες σας, απόψεις, ιδέες. Θέλουμε τις απόψεις σας για να αναπτύξουμε περαιτέρω τη μεθοδολογία μας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας και την επικοδομητική συνεισφορά σας σε αυτή την ε, σημαντική προσπάθεια και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Θα δώσουμε το λόγο στον συγητή, στους συγητές. Δεν είναι εδώ και ο Σκάρενς. Η κυρία Σαρτζεντίνη έχει το λόγο που είναι εισηγήτρια την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Τιμή μου, κύριε Πρόεδρε. Ε, όχι, δεν εννοούσα ότι είστε δεύτερη επιλογή. Ε, ενώ, εντάξει, η ΕΚΟΝ προηγείται. Μα το ήξερα, ήξερα τι θα πείτε. Και όμως δεν μπορείτε, γιατί εγώ τα έχω συμφωνήσει εδώ με τον συνάδελφο τον Πράσινο για το ποιο θα μιλήσει. Ε, μα εγώ δεν το ήξερα, λέει ο Πρόεδρος. Τι λέγατε με τον κύριο Γκίγκολντ. Οπότε θα περιμένω να έρθει η σειρά των πρασίνων και με συγχωρείτε. Ε, δεν μπορώ να προβλέψω και τι θα κάνουν οι πράσινοι, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Γκίγκολτ, θα μιλήσετε εξ του κύριου Κάρινς. Ε, δεν ξέρω τώρα εάν είναι σωστό αυτό και αν θα χαιρόταν ο κύριος Κάρινς, αν και υπάρχει βεβαίως κάποια προσέγγιση μεταξύ των δύο ομάδων μας. Ε, τέλος πάντων τώρα μην μπούμε στις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Ας ε, πάμε με τη σειρά, ας ακούσουμε το ΕΛΚ ε, και το πώς θα καταπολεμήσει το ξέπλυμα του χρήματος. Α, και τελικά θα μιλήσω εγώ, λοιπόν. Εγώ ήθελα απλά να μιλήσει ο εισηγητής της Λίμπε πρώτος. Θα μιλήσετε λοιπόν εσείς εξ ονόματος του κυρίου Κάρενς. Όχι, όχι, κάποια γενικά σχόλια θα έκανα. Μπορούμε να ακούσουμε πρώτα τους συνεισηγητές. Λοιπόν, Σαρτζεντίνη και μετά θα περάσουμε στου υπόλοιπου ομιλητέ. Εντάξει, μα δεν κάνω, δεν, δεν έκανα, δεν αστευόμουν. Τέλο πάντων, να πω δύο λόγια έτσι αφού επιμένετε. Νομίζω ότι είναι δεκτέ οι εξηγήσει τη Επιτρόπου. Είναι μακρά η πορεία. Έχουμε πει δύο φορέ όχι σε πράξη κατεξοδότηση. Εν τω μεταξύ συνέβησαν κάποια πράγματα έτσι, και πολλά έχουν αλλάξει προ το καλύτερο και το γεγονός ότι βεβαίως προτείνατε μία λίστα με κριτήρια είναι αιτία αισιοδοξία για όλους μας. Λοιπόν, θα αφήσω τις λεπτομέρειες για να τις πει ο συνάδελφος μετά. Ευχαριστώ. Μάλιστα, κανένας άλλος δεν έχει ζητήσει το λόγο. Αυτό είναι το άλλο πρόβλημα. Πέρα από τον κύριο Γκίγκολτ, ποιος άλλος είναι στον κατάλογο των ομιλητών. Okay, who, who else is on the list? On the list. Uh, Λοιπόν, μάλιστα, κύριε Γκίγκολτ. Uh, funnily um, η κυρία Μετσόλα και ο κύριο Γκίγκολτ είναι στον κατάλογο των ομιλητών. Ποιο θα μιλήσει τελικά. Μα ο ένα παραχωρεί το βήμα στον άλλον. Λοιπόν, ωραία, θα ξεκινήσω εγώ. με έχουν μπερδέψει όλα αυτά. Ευχαριστώ, εν περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την Κομισιόν για τις ε, εξηγήσει που βασίζονται στον οδικό χάρτη που μας παρουσιάσατε ήδη και οφείλω να πω ότι θεωρώ ότι αυτά τα κριτήρια και οι προτεραιότητες μου φαίνονται λογικές και λογικά. Μία ερώτηση έχω μόνο για τα κριτήρια χωρών που ίσως κατονομάσει η Europol. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος τρόπος να συλλέξουμε δεδομένα από εθνικές περιπτώσεις για το ποιες τρίτες χώρες ε, εμφανίζονται τακτικά στα δικαστήρια για περιπτώσεις ξεπλήματος χρήματος για να έχουμε έτσι κάποια αντικειμενικά δεδομένα που παράγει ούτως ή άλλως ε, το νομικό μας σύστημα και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια αφετηρία για να δούμε ποιες χώρες είναι ε, προβληματικές. Υποψιάζουμε ότι η Αιθιοπία και οι Λιπές ε, μάλλον σπάνια θα εμφανίζονται. Αλλά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια καλή πηγή πληροφοριών και για τη δικιά σας τη δουλειά. Τούτου λεχθέντος. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο ζητήματα που ετέθησαν εδώ στην προηγούμενη συνεδρίαση όταν δυστυχώς λείπατε και χαιρόμαστε τέλος πάντων που έχετε αναρρώσει. Πρώτα απ' όλα η προθεσμία για το 2025. Καλό θα ήταν να ξέρουμε πότε θα έχουμε έναν πρώτο γύρο και ε, ιδεώδες θα ήταν ε, βεβαίως ε, να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος πριν από το 2025. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο ετέθη από αρκετούς συναδέλφους, είναι το θέμα της στελέχωσης. Έχουμε δει την αύξηση του προϋπολογισμού στην ε, ομάδα εργασίας αυτήν για το οικονομικό έγκλημα, αλλά δεν αρκεί. Οπότε, αν το συγκρίνουμε με τις ΙΠΑ και το ότι επενδύουν ε, στην καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος, ε, εντάξει, είναι δυσανάλογο, δεν είμαστε ΙΠΑ, αλλά παρά είναι δυσανάλογο. Ε, είναι, έχουν ε, τριψήφιο αριθμό ατόμων που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Οπότε οι ΙΠΑ συχνά είναι πιο σκληρές σε διεθνές επίπεδο για αυτά τα ζητήματα και δεν προξενεί έκπληξη. Οπότε εγώ θα το εκτιμούσα αν υπήρχε κάποια περαιτέρω δέσμευση όπως έκανε ο κύριος Γιούνκερ στην ε, συνεδρίασή μας, στην ακρόαση μας. Δηλαδή δύο θέσεις δεν αρκούν. Και ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε να κάνει ένα οργανόγραμμα και να μας πει πόσα άτομα θεωρούν ότι χρειάζονται για αυτή τη δουλειά. Οπότε έχουμε και ευθύνη και ως εργοδότες και οι άνθρωποι αυτοί πόσο να δουλέψουν δηλαδή, δεν μπορεί να κοιμούνται και μες στο γραφείο και οι σοσιαλδημοκράτες και άλλοι θα έχουμε κάποιες ανησυχίες αν δεν μπορούμε να συμβαστούμε κάποια όρια στο ωράριο αυτών των ανθρώπων. Κάποιοι, άνθρωποι, βέβαια, κάποιοι συνάδελφοι είναι κατά της ε, σχετικής οδηγίας, αλλά ε, πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να μην πάθουν υπερκόπωση. Και τέλος, ε, μια εμπειρία από τη Μάλτα. Η FATF και η πρόσφατη επίσκεψή μας ως αντιπροσωπεία των Επιτροπών Λίμπε και Πάνα έχουμε Αζερβαϊτζάν, για το οποίο ξέρουμε ότι είχαμε κάποιες περίεργες ροές και στη Γερμανική Βουλή έφτασε το θέμα. Δεν είναι στη λίστα FATF. Γνωρίζουμε πολλές περιπτώσεις πολιτικής επιρροής με αζέρικα χρήματα αλλά δεν είναι στην λίστα του FATF. Θα πρότεινα λοιπόν να ρίξετε μία ματιά εκεί γιατί μάθαμε στη Μάλτα ότι επειδή το κεφάλαιο έρχεται σε μία, από μια τράπεζα αζερική δεν είναι αυτό από μόνο του λόγος ανησυχία. Αυτό είναι κάπως προβληματικό. Και ξέρουμε και την δύσκολη κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε σας ευχαριστώ για τις κινήσεις που κάνατε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πάσχα, το οποίο νομίζω μπορεί να αποτελέσει ένα σύμβολο για την δύναμη της Ευρώπης όταν δράει ενωμένη. Κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ πολύ, Κλώτ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όπως και στα αδελφή μου εσάς, κύριε Επίτροπε, που ήρθατε εδώ και κάνετε τόσο πλήρη παρουσίαση του, του χρονοδιογράμματος και του προγράμματος εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το ότι καταλήξαμε επιτέλους σε μία μεθοδολογία θα είχαμε προτιμήσει όμως να ήμασταν και λίγο περισσότερο φιλόδοξοι. Δεν ξέρω αν μπορούμε κάπως να επιταχύνουμε την όλη διαδικασία. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 2025 και εσείς το είπατε εσείς, αλλά νομίζω ότι οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα έχει στο πότερο στόχο του 2025 θα πρέπει ουσιαστικά να τροποποιηθεί προκειμένου να γίνει λίγο πιο φιλόδοξο και να επιταχυνθεί τροποντινά. Αν αυτό σημαίνει θα πρέπει να προβληθεί πιο ενισχυμένο προσωπικό, τότε εμεί ω πολιτική ομάδα σαφώ το προτιμάμε. Πέρα από αυτό, το ΕΛΚ αλλά και εγώ προσωπικά ως Ευρωβουλευτής από τη Μάλτα θα συμφωνήσω μετά σου είπε ο κύριος Γκίγκολτ για το Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε τώρα να καλύψουμε όπως βλέπετε όλες τις πολιτικές ομάδες. Από τους σοσιαλιστές υπάρχει κάποιος που θέλει να πάρει το λόγο. Η το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για το ότι τηρήσατε την δέσμευσή σας. Μολόν καταλαβαίνω ότι κάποιοι λόγοι πέραν από το δικό σας τον έλεγχο σας ανάγκασαν να αναβάλλετε την αρχικά προγραμματισμένη συνάντησή μας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα πλαίσια μιας διαδικασίας που ξεκινήσει εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο δικός χάρτης μας προτείνεται, συνάδει πλέον με ζητήματα τα οποία έχουμε θίξει εμείς στο παρελθόν, Ωστόσο αναφερθήκατε πολύ στο ότι θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, αλλά είπατε ότι αυτό εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου όσον αφορά την οδηγία για την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων παράνομες δραστηριότητες. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα πρέπει να λάβει όντω χώρα, αλλά υπάρχουν και κάποια κριτήρια τα οποία δεν εξαρτώνται από την διαπραγμάτευση αυτή. Επομένω, θα πρέπει και εσεί ω Επίτροπο, γενικότερα ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μπορείτε να λάβετε και αυτόνομα δάση. Δεν ξέρω αν από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, σε σχέση με τα κριτήρια αυτά, έχετε καταφέρει να σημειώσετε μια κάποια πρόοδο, να μας πείτε ποια είναι τα κριτήρια αυτά και δυνατόν ήδη από σήμερα να ενημερωθούμε για αυτά. Πέρα από αυτό, αναγνωρίστε και εσείς ότι θα πρέπει η Ευρώπη να μπορεί να κινηθεί αυτόνομα σε σχέση με άλλους οργανισμούς όπως η ομάδα ΓΚΑΦ, η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης. Βλέπετε όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη παγκόσμια συνειδητοποίηση η οποία απορρέει από τα Paradise Papers ή από άλλες εργασίες που, που γίνονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι οποίες επηρεάζουν τελικά την κατάρτιση, την εκπόνηση αυτών των καταλόγων. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να είμαι όντως βέβαιη ότι η νέα αυτή μέθοδος μας προτείνεται δεν θα μας οδηγήσει απλώς στο να ακολουθούμε εμείς τις δραστηριότητες και τις εξελίξεις στα πλαίσια του γκάφη, ερχόμενη βέβαια σε δεύτερη θέση. Και αν δείξετε υπέρμετρη εμπιστοσύνη στο Συμβούλιο, δεν νομίζω ότι θα καταφέρετε να σημειώσετε πρόοδο. Ποιες διασφαλίσεις μας δίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να μην καταλήξουμε σε ένα διέξοδο, να είμαστε δέσμοι τελικά των αποφάσεων του Συμβουλίου. Και κάτι τελευταίο και απευθύνομαι και στον Πρόεδρο. Γίνεται συζήτηση σήμερα το βράδυ. Ακούσαμε έναν οδικό, στην οδικό χάρτη που υπάρχει ήδη από τον Ιούνιο. Από νομική πλευρά όμω δεν μα παρουσιάζεται τίποτα το απτό. Πέρα από όλα αυτά λοιπόν Μήπως θα έπρεπε να έχουμε μια ανταλλαγή επιστολών ή κάτι ακόμα, κάτι διαφορετικό, προκειμένου πραγματικά να δούμε ποια είναι η έμπρακτη δέσμευσή σας σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, πέρα από την ολοκλήρωση πραγματεύσεων για την οδηγία AMLD, θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποιες άλλες δεσμεύσεις αναλαμβάνετε εσείς. Γιατί δεν εξαρτώνται τα πάντα από την εκπόνηση των κριτηρίων εκείνων στα πλαίσια της οδηγίας AMLD. Πρέπει να έχουμε και άλλες δεσμεύσεις από εσά, Πρόεδρος. Πρέπει να ολοκληρώσουμε πριν τις 7.30, λέει ο Πρόεδρος, και πρέπει να ψηφίσουμε ενδεχομένω εν συνεχεία. Εξ ονόματος TCR δεν θέλει να πάρει κανείς το λόγο, από ό,τι βλέπω. Ο κύριος Τζέζεκ τώρα από τους φιλελεύθερους. Δύο με τρία λεπτά το πολύ, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Προχωρήσαμε αρκετά. Ερώτηση έχω για τα κριτήρια. Εδώ καθορίζουμε άλλα κριτήρια στο χάρτη πορείας, πέρα από την οδηγία. Εν ώψη τριμερούς διαλόγου, ποια είναι η άποψη για τη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία, του του πραγματικό ιδιοκτήτη μιας εταιρεία. Ευχαριστώ. Για τους πρασίνους. ΕΝΕΦ. Γκουε. Όχι. Ο κύριος Βιέρας. Δύο-τρία λεπτά. Δεν και ο ηγετής αλλά παρόλα αυτά, εν συντομία, έχω να πω κάποια πράγματα. Βέβαια, δηλώνουμε τα προφανή εδώ. Δεν ικανοποιεί αυτό ούτε στο ελάχιστο τις θεμητές προσδοκίες των πολιτών. Πόρο απέχει από την αντιμετώπιση των ευθυνών που απορρέουν από σειρά σκανδάλων. Χρειάζεται πιο καλή, πιο στοχευμένη δράση. Αυτή είναι η άποψή μας. Ο κατάλογος δεν αλλάζει ουσιαστικά. Ούτε καν σε σχέση με δημόσιες εκδηλώσεις. Μια προσπάθεια για προσθήκη κριτηρίων δεν μπορούμε να αντιγράφουμε παλαιότερους καταλόγους. Το αποτέλεσμα υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών. Και αν κινούμεθα θα πλήρη κατάλογο το 2025, πώς θα δικαιολογηθούμε για την καθυστέρηση στους πολίτες μας. Είναι απαράδεκτο κατά την άποψή μου. Δεν είναι ερώτηση αυτή. Αυτή είναι η αρχική μου εντύπωση. Ο κ. Κόμπερν για το EFTD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να μιλήσω και για το συναλλαγματικό έλεγχο. Τροπολογία Α για τους νομισματικούς ελέγχους. Η βασικά αγαθά, δηλαδή αγαθά υψηλής, υψηλότερης αξίας σε σχέση με το μέγεθός τους. Αυτό τι είναι για το επόμενο σημείο. Άλλο θέμα, άλλο θέμα. Α, μετά αυτό. Δεν έχει νόημα. Ε, είναι λογικό, αλλά δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε τώρα αργότερα. Αργότερα είναι η απάντηση, λέει και ο Πρόεδρος. Κύριε Σάιμον, ο τελευταίος ομιλητής. Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να επαναλάβω ένα ερώτημα του κυρίου Γκίγκολτ που είχα και εγώ. Το θέμα του προσωπικού. Θυμάμαι τα επιχειρήματα της Κομισιόν στην αρχή για το πόσο χρειάζεται, πόσο καιρό χρειάζεται για να ερευνήσει κάποιες χώρες και να ε, καταρτήσει μια τέτοια λίστα. Και βεβαίω ε, δεν μπορεί να είναι πάρεργο κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένα λοιπόν το ερώτημα του κυρίου Γκίγκολτ. Πόσες θέσεις ισοδύναμες πλήρους απασχόλησης θα υπάρξουν περισσότερες από όσους είχαμε στο παρελθόν. Αλλιώς δεν γίνεται να συντάξουμε μια τέτοια λίστα. Μια δεύτερη ερώτηση. Πρέπει στο μέλλον να αποφύγουμε το να ξαναβρεθούμε στη θέση που ήμασταν στους τελευταίους μήνες. Δηλαδή, να καταλήξουμε κάπου, να ολοκληρωθεί η εργασία μας και μετά βεβαίως να μην γίνεται δεκτή. Όταν θα συντάσσουμε λίστες στο μέλλον θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πριν οριστικοποιηθεί η πρότασή σας δηλαδή να υπάρξει μια συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακριβώς για να αποφύγουμε αυτά τα οποία είχαμε και να καταλήγουμε σε κάποιες ε, προτάσεις καταλόγων που θα δέχεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πίτερ, να δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Επίτροπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από το τέλος, ε, το σχόλιο των κυρίων Σίμων και Γκίγκολ για τις ε, δυνατότητες. Θα χρειαστούμε επαρκείς δυνατότητες για να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις ε, που ε, ανοιχτά είπα ότι αναλαμβάνουμε. Έχουμε ήδη ενισχύσει την στελέχωση της ε, σχετικής μονάδας, μιας καινούριας μονάδας που συστήθηκε για τον σκοπό αυτό και θα αναδιοργανώσουμε τις ικανότητες και το προσωπικό εντός της Γενικής Διεύθυνσης ε, για να καταλήξουμε σε έναν κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου μέχρι το τέλος του 2018. Χαίρομαι που έχω τη στήριξη του Κοινοβουλίου αλλά και του Ζαν Κλοντιούνκερ που είπε σαφώς ότι αν υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί το προσωπικό θα δώσει το πράσινο φως. Πρέπει να πω κάτι ακόμα. Αυξάνοντα ε, το προσωπικό επίσης ε, μιλάμε και για προσωπικό από τα κράτη-μέλη. Άκουσα εδώ πέρα το σχόλιο ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τα κράτη-μέλη. Εγώ εμπιστεύομαι τους ειδικού που συνεργάζονται μαζί μας και θεωρώ ότι δημιουργώντας ένα κοινό περιβάλλον εργασίας και ένα κοινό καθεστώς εργασίας θα καταφέρουμε να κάνουμε την δουλειά μας. Βεβαίω, πρώτα απ' όλα είναι η ευθύνη της Κομισιόν, ευθύνη την οποία αναλαμβάνω πλήρως και με κάθε σοβαρότητα. Σας λέω ότι θα υπάρχει η απαραίτητη στελέχωση. Τώρα για να επανέλθω στα σχόλια και τις ερωτήσεις ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σαρτζεντίνη για την αισιοδοξία της. Κύριε Γκίγκολ τώρα, ποιες είναι οι πηγές πληροφοριών και τι μορφή θα έχουν οι πληροφορίες που δίνει η Europol. Βεβαίως για ευνόητους λόγους ε, θα περιληφθεί και η Europol γιατί έχουν ε, διάφορες πληροφορίες ε, από πολλές πηγές ε, και από τις εθνικές υποθέσεις όχι μόνο όσε καταλήγουν στα δικαστήρια, αλλά και πριν από αυτή τη φάση. Έχουν τις πληροφορίες από τα κράτη-μέλη και τις πηγές ε, που τους δίνουν πληροφορίες για τρίτες χώρες. Οπότε, λογικά, σκεπτόμενοι, καταρτίζοντας αυτήν την λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ε, τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, θα χρησιμοποιήσουμε ακριβώς αυτούς τους διάβλους ε, και τις πληροφορίες της ε, Europol. Βεβαίως υπάρχουν κάποια όρια στο τι πληροφορίες μπορούν να δώσουν τα κράτη-μέλη, αλλά τέλος πάντων ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Για την ε, προθεσμία 2025 και τι θα γίνει μέχρι τότε. Κοιτάξτε, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους υποσχέθηκα να εγκρίνουμε τον κατάλογο. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο έτος, με βάση αυτήν την μεθοδολογία, θα έχουμε την αξιολόγηση των χωρών που θα αξιολογηθούν. Και βεβαίως εντωμεταξύ πρέπει να εργαστούμε με τις πληροφορίες που έχουμε για το λεγόμενο αζέρικο πλυντήριο. Όχι μόνο για τις χώρες όπου υπάρχει δηλαδή η υποψία ότι κάτι τρέχει, αλλά υπάρχουν και κάποια προβλήματα ad hoc. Γι' αυτό ακριβώς ε, έχουμε και αυτό το χειρόφρενο. Οπότε θα λάβετε του χρόνου τις πληροφορίες για τον πρώτο γύρο αξιολόγησης με την δυνατότητα να προσθεθούν και άλλες χώρες ανά πάσα στιγμή. ο κατάλογος θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 18 και θα συνεχιστεί η δουλειά, θα προστίθενται δηλαδή νέες χώρες σύν χρόνο μέχρι το 2025. Είπα και πριν ότι χρειάζεται η μέγιστη δυνατή διαφάνεια εδώ. Οπότε τα κράτη-μέλη τα οποία συνεργάζονται στο θέμα αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ενήμερα για κάθε βήμα που κάνουμε. Οπότε τώρα δεν μπορώ να σας πω ποιο μήνα ακριβώς του 18 θα έχουμε τον πρώτο κατάλογο των χωρών προς αξιολόγηση, αλλά δεν θα είναι Δεκέμβριο κάποια στιγμή και θα προσπαθήσουμε να είναι το στομότερο δυνατόν. Για το Αζερβαϊτζάν μίλησα και εκτιμώ ότι θα είναι μεταξύ των χωρών αυτών που θα αξιολογηθούν. Κύρια Μετσόλα, ναι, μιλήσατε για μεγαλύτερη φιλοδοξία, περισσότερο προσωπικό, Αζερβαϊτζάν, ναι, τα απάντησα αυτά. Κυρία Μπερές, είχαμε μακροσκυλής συζητήσεις ε, και ξεκαθάρισα ότι πρέπει να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Διακυβεύονται πολλά πράγματα, όχι μόνο η σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος ή η μακροοικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η ίδια η εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα λοιπόν. και οπωσδήποτε θα υιοθετήσουμε την αναλογή μεθοδολογία και με το κατάλληλο προσωπικό θα τα καταφέρουμε. Κύριε Γεζακ, ε, εγώ είμαι ανοιχτή σε μια θετική προσέγγιση για την διεύρυνση του άρθρου 9 στην οδηγία περί ξεπλήματος χρήματος. Είχα πει και την άλλη φορά ότι η διαφάνεια για μένα είναι ένα από τα κύρια κριτήρια. Αυτή είναι, θα έλεγα, η θετική μου αντίδραση. Για να δούμε το πώς θα συνεχιστεί η υπόθεση αυτή στον τρίμερη διάλογο, που ελπίζω να γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβουργό, για από τους πράσινους τώρα. Λοιπόν, δέχομαι την κριτική που μου ασκήσατε και απαντώ ότι είμαι πεπισμένη ότι η προτινόμενη από εμά μεθοδολογία είναι η καλύτερη δυνατή. Αν εσεί έχετε να κάνετε κάποιε προτάσει βελτιωτικέ, ε, ή αν έχετε να προτείνετε μια διαφορετική προσέγγιση, Εμεί είμαστε πολύ διαλλακτικοί και με ανοιχτό πνεύμα θα ακούσουμε τι προτάσει σα. Θεωρώ πάντω ότι προτείνουμε ένα σύστημα το οποίο έχει μια στρατηγική συστηματική προσέγγιση με ad hoc ε, επιτόπου γρήγορες αντιδράσεις όταν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες. Αυτή είναι λοιπόν η απάντηση που είχα να σας δώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Απευθύνομαι στους συντονιστές. Προτού προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Θέλετε να κάνουμε μεταξύ μόνο κάποια συζήτηση για την μήνυ αυτή ακρόση που είχαμε όχι από τους φιλελευθέρους και από κανέναν άλλον. Ακούσαμε λοιπόν την Επίτροπο η οποία μας παρουσίασε τη μεθοδολογία της να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου είναι προθεσμία για να εκφράσουμε αντίρρηση. Αν εκφράσουμε αντίρρηση θα πρέπει αυτή να ψηφιστεί στην Ορομέλεια του Δεκεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε την απλουστευμένη διαδικασία αν να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο ψηφίσματος αντίρρησης και θα πρέπει βέβαια να συμφωνήσουν επ' αυτού και οι συντονιστές. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν υπάρχει αντίρρηση Κύριε Επίτροπε, σε ευχαριστούμε για την συμβολή σας σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να μας συναντήσετε, ενώ σας το ζητήσαμε τόσο τελευταία στιγμή και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε στην Επιτροπή μας πολύ σύντομα.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 Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf nochmals, weil Λοιπόν, μια που έχουμε τόσου πολλούς ε, συναδέλφου που ήρθαν τώρα, σα καλωσορίζω στην κοινή μα ε, συνεδρίαση των Επιτροπών ΛΥΜΠΕ και ΕΚΟΝ, όπου τώρα θα ασχοληθούμε με την ψηφοφορία της έκθεσης Ντελβό και Ακογιάρ για τους ελέγχους ε, στις χρηματικές ροές. Ελπίζω να είναι καλή η ε, ψηφοφορία. Για μένα θα είναι η πρώτη σε αυτόν τον ρόλο. Να βάλω τα γελιά μου να σας βλέπω. Ευχαριστώ τους εισηγητές για τις συμβαστικές προτάσεις. Γίνονται έτσι τα πράγματα απλούστερα. Πρώτα απ' όλα θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Εγώ δεν έχω κάρτα, κάποια στιγμή θα μου τη φέρουν. Κάπου εκεί είναι τώρα, αλλά... Κάπου την πήρανε, την τακτοποίησαν στο ενδιάμεσο. Λοιπόν, δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Ναι, ναι μετά, μετά, τώρα. Να δούμε αν δουλεύουν τα μηχανήματα. Πάμε. πέρας και... Όλοι εδώ. Ωραία. Πριν περάσουμε στην πραγματική ψηφοφορία, να δώσω τον λόγο στον συνεισηγητή, τον κύριο Χουάν Φερνάντο Λόπεζ Αγγιγέρ. Είναι θυμικό δίκαιο να ευχαριστούμε όλους, κυρίως τους σκιώδεις, για το νομοθέτημα. Λυπούμε που η κυρία Ντελβό απουσιάζει ως συνεισηγήτρια. Να πω σε όλους ότι προσπαθήσαμε να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία με αυτό το εργαλείο που έχει στόχο μέσω εσωτερική αγοράς θέλει να ενισχύσει τον έλεγχο το διασυνοριακού μετρητού Σε εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διαφυλάσσοντας όμως τα θεμητά συμφέροντα Άρα αναλογική προσέγγιση. Και εξασφαλίσαμε ότι θα υπάρχει και ρήτρα αναθεώρησης, όπως αποκαλείται. Κάθε τρία χρόνια για να μπορεί να μαθαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να βελτιώνει το νομοθέτημα που πρόκειται να υιοθετήσουμε. Ευχαριστώ. Chairman. Vielen Dank für diese Einführung. ευχαριστώ για την εισαγωγή αυτή. Τι γίνεται. Να. Κάποιος πάλι θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Πού είναι. Ναι, κύριε Κόμπερν. Um, Πρόεδρε, φρικάρισα από το συμβιβασμό Α. Αντιβαίνει τα πάντα υποχρέωση για δήλωση προσωρινών λεπτομεριών, το αποστολέα και το αποδέκτη και προέλευση και πρόθεση χρήσεως των μετρητών. Περιορισμό τη έκφραση πρώτα απ' όλα, διότι τα χρήματα μιλούν, άρθρο 10 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, άρθρο 8 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Απαγορεύει και όλο τον περιορισμό ε, μάλλον περιορισμό, περιορίζει την ε, μεταφορά χρημάτων. Άρθρο λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ασταδιακά να καταργήσει τις απαγορεύσεις στο διεθνές εμπόριο. Ναι, να, να σας διακόψω κύριε Κόμπερν. Είναι περιορισμός της ελευθερίας του κεφαλαίου και είναι ασφαλμένο. Θυμίζει τον έλεγχο συναλλαγματο του δεκαετίας του 70, το είχαμε στη Βρετανία, που μπορούσες να βγάλεις ναι, μόνο 50 λίρες, ήταν καταστροφικό. Έπρεπε να μάθω. Μάλιστα τώρα βρήκα το κουμπί, ωραία κύριε Κόμπερν. Οι συμβαστικές εδώ πέρα συμφωνήθηκαν μεταξύ των ε, εισηγητών, με τους σκιώδεις εισηγητές και έτσι συμφώνησαν. Ειλικρινά, λυπούμε αν δεν σας αρέσουν, έτσι είναι όμως οι κανόνες και τώρα ψηφίζουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε την τροπολογία 81 της κυρίας Κάπελ. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, όχι ηλεκτρονική, όχι. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Άρθρο 137. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική αλφα. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική β. Υπέρ κατά δεκτή 32 υπέρ κατά δεκτή συμβαστική C υπέρ κατά δεκτή 165 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε Ψήφισαν, έχουν όλες τις κάρτες εκτός μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Συν ένας υπέρ εγώ δεκτή. Συμβαστική D υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 176 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 47 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική F υπέρ. Κατά. Δεκτή. Α, όχι. 51 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 186 υπέρ. Κατά. Α, απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 187 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική G υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική H υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική I υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική J υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική K. Αφού έτσι θέλετε. πρέπει να εγώ νομίζω ήταν σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Συν Ένα εγώ υπέρ πέρας και 32 υπέρ 27 κατά δεκτή συμβαστική που ήμασταν κάπα υπέρ κατά δεκτή 210 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική L υπέρ κατά δεκτή 67 υπέρ κατά δεκτή 213 αποσύρεται συμβαστική M υπέρ κατά δεκτή συμβαστική N υπέρ κατά δεκτή 216 υπέρ κατά δεκτή συμβαστική όμικρον υπέρ κατά δεκτή συμβαστική π υπέρ κατά δεκτή 228 υπέρ κατά απορρίπτεται 229 μέχρι 235 όλες μαζί 229 μέχρι 235 unblock υπέρ κατά απορρίπτεται 230 υπέρ όπα όχι μια στιγμή υπέρ κατά όχι όχι 73 73 συγγνώμη 73 υπέρ κατά δεκτή 74 υπέρ κατά δεκτή 75 υπέρ κατά δεκτή 243 υπέρ κατά απορρίπτεται 244 υπέρ κατά δεκτή 245 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε με την κάρτα μου επιτέλους άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 246 υπέρ κατά δεκτή συμβαστική Q υπέρ κατά δεκτή 79 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 251 υπέρ. Απορρίπτεται. 254 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 255 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 256 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 257 υπέρ. Και 58 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 259 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 260 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στις ε, αιτιολογικές αναφορές. 1 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 83 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. να την ξαναδούμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και... Εγκρίνεται. Και είμαστε 85 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 1. Όχι 86 υπέρ. Κατά. Ναι, ναι, ναι. Δεκτή. 87 υπέρ. Κατά. Δεν θέλω και αυτή να τη δω. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, ναι, όχι, ήταν σαφές. 88 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 89 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 91 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 3. 4. 96 και τα λοιπά. Για να δούμε. Κάτι δεν, δεν πάει καλά. Λοιπόν, τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 96 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική R υπέρ. Κατά. Δεκτή. 106 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 107 αποσύρεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 108 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά δεκτή. 8 υπέρ κατά δεκτή. 109 υπέρ κατά απορρίπτεται. 110 υπέρ όχι 111 μαζί υπέρ κατά απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά δεκτή συμβαστική S υπέρ κατά α, δεκτή 114 υπέρ κατά δεκτή 116 υπέρ κατά απορρίπτεται 117 υπέρ κατά απορρίπτεται 118 υπέρ κατά απορρίπτεται 119 υπέρ κατά απορρίπτεται 11 υπέρ κατά δεκτή 122 υπέρ κατά δεκτή 12 υπέρ 124 υπέρ κατά απορρίπτονται 123 υπέρ κατά δεκτή 13 υπέρ κατά δεκτή 14 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 15 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 125 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ταφ υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 18 ε, υπέρ. Κατά. Δεκτή. 129 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 130 υπέρ κατά δεκτή 131 υπέρ ορίστε ε, συμβαστική U υπέρ κατά δεκτή 133 υπέρ κατά απορρίπτεται 134 υπέρ κατά απορρίπτεται 21 υπέρ κατά δεκτή συμβαστική β υπέρ κατά δεκτή εκτιμώντα 136 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται λοιπόν ψηφίζουμε τώρα την πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία υπέρ Ποιος? Μάλιστα, πέρας. Σαφής πλειοψηφία. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 80 το νομοθετικό ψήφισμα ε, χωρίς όμως υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Οπότε και τέλος ψηφίζουμε την απόφαση να πάμε στις διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση την έκθεση που εγκρίναμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Οπότε μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ και καλό σας βράδυ. Λίγα τη συνεδρία.